Ε, η παρέμβαση για διαδικαστικό θα λάβει αμέσως τον λόγο κύριε Γκλέσο. Η Επιτροπή Μεταφορών έχει ένα διορθωτικό σε σχέση με ένα κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 231 εδάφιο 4. <clears throat> Αυτό το διορθωτικό θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται αν μέχρι 20, μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωσή του δεν δηλωθεί από 40 μέλη ότι πρόκειται να ψηφιστεί προς έγκριση. Και έτσι λοιπόν ο τίτλος θα αναφέρεται στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασής μας. Μετά από τη διακοπή της περίοδου συνόδου